δηλαδή εις ε, τον κοινό προγραμματισμό σχετικά με ε, τις ψυχικές ασθένειες και ιδίως το Αλτσχάιμαρ. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ρόιλ, ο οποίος έχει καθυστερήσει και μας είχε πει εκ προημίου ότι θα καθυστερήσει γι' αυτό και προτείνω να ακούσουμε καταρχήν την κυρία Γκροστέτ και στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Η κυρία Γκροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, δεν είναι εδώ ο κύριος Ρόιλ Οπότε εγώ θα υπενθυμίσω την ερώτηση αυτή που θέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της νομικής ε, βάσης άρθρο 165 της Συνθήκης. Πρόκειται για σύσταση του Συμβουλίου για μέτρα καταπολέμησης των ευρωεκφυλιστικών νοσημάτων. Ζητάμε Μάλλον χρειάζεται να γίνει διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Αυτό απαιτεί η νομική βάση. Το Συμβούλιο λοιπόν ρωτάω μπορεί να επιβεβαιώσει την ε, θέση του ότι θα περάσει στις 3 Δεκεμβρίου 2009 στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού το θέμα αυτό. Και εφόσον υπάρχει διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα λάβει υπόψη του την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταλήξει όσον αφορά το θέμα αυτό. Επίσης, όταν θα έχουμε αργότερα πρωτοβουλίες για προγραμματισμό από κοινού των ερευνητικών δραστηριοτήτων, το Συμβούλιο μπορεί να μας επιβεβαιώσει τη γνώμη του ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει καταρχήν να εγκριθούν όλες με την ίδια νομική βάση. Υπενθυμίζω εδώ ότι έχουμε συντάξει ψήφισμα. Το ψήφισμα αυτό συμπεριλαμβάνει τη συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων. Και είναι σημαντικό αυτό το ψήφισμα γιατί απλά μιλάει για την γύρανση του πληθυσμού και το τι διακυδεύεται εξαιτία αυτή τη ε, γύρανση. Έχουμε πάνω από 7 εκατομμύρια που πάσχουν από Αλσχάιμερ στην Ευρώπη σήμερα και σύμφωνα με τι προβλέψει θα διπλασιαστεί το νούμερο αυτό μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επενδύσουμε, να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα ώστε να ελέγξουμε το κοινωνικό κόστο, να δημιουργήσουμε ελπίδα, αξιοπρέπεια στα εκατομμύρια ανθρώπων που πάσχουν από Αλσχάιμερ. Τα, ζητήματα αυτά των ε, νευροεκφυλιστικών νοσημάτων αφορούν την κοινωνία, αλλά την κοινωνία σε όλες τις ευρωπαϊκές ναι. χώρες. Χρειάζεται λοιπόν διάγνωση, χρειάζεται θεραπεία, φάρμακα. Πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε τη στήριξη λοιπόν στην έρευνα και στην ε, καινοτομία με συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για να βρούμε νέε θεραπείε και να αντιμετωπιστούν τα νοσήματα αυτά. Η έρευνα στον τομέα τη έρευνα είναι πολύ κατακαιρματισμένη ακόμα μέσα στην Ευρώπη και η εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα πρέπει να πολλαπλασιαστεί. Χρειαζόμαστε νέα φάρμακα. Η σχετική δίωξη ξεκίνησε τον ε, Φεβρουάριο. Πρέπει να συνεχιστεί. Πρόκειται για έναν ε, αγώνα που κάνουμε κατά του χρόνου. Υπάρχουν τρόποι για να γίνεται έγκαιρα διάγνωση. Είναι λοιπόν αυτά τα συγκεκριμένα θέματα για τα οποία οι πολίτες περιμένουν ένα μήνυμα από την Ευρώπη, περιμένουν κάποιες εγγυήσεις ώστε να μπορέσουν να προλάβουν νοσήματα τέτοια που έχουν να κάνουν με τη γύρανση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Γκροστέτ. Ε, για πέντε λεπτά έχει το λόγο η κυρία Μάλστραμ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η πρόταση για μία σύσταση του Συμβουλίου για τα μέτρα ε, σχετικά με το Alzheimer υιοθετήθηκε 22 Ιουλίου εφέτος και βασίζεται στο άρθρο 165 στο Συμβούλιο κατά τρόπον ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για τεχνολογικές εξελίξεις και για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει καλύτερο συντονισμός της εργασίας η οποία γίνεται. Το άρθρο 165 ε, και η πρωτοβουλία για κοινό προγραμματισμό ε, αλληλοσυμπληρώνονται και με τη βοήθεια των κρατών μελών μπορέσαμε να κατατήσουμε καλά κοινά προγράμματα με στόχο να, αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, της χρηματοδότησης της δημοσίας έρευνας στην Ευρώπη. Το άρθρο αυτό δεν δίνει στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να δράσει αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μεταξύ των κρατών μελών και του Συμβουλίου γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταρτιστεί κοινό προγραμματισμός. Υπάρχει πολιτική βούληση του Συμβουλίου να προωθήσει τις πρωτοβουλίες για κοινό προγραμματισμό και να καταπολεμήσει αρρώστιες σαν το Αλτσχάιμερ το ταχύτερο δυνατόν. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του Συμβουλίου θα πρέπει να υιοθετηθούν προτάσεις βάσει του κειμένου που έχει προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση του Αλτσχάιμερ και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησαν από το καλοκαίρι ότι αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος για τη δημόσια ιδέα εξού και αυτή η πρόταση πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Προεδρία θα μπορέσει να λάβει υπόψη αυτά τα οποία είπε το Συμβούλιο όταν καταλήξει στα συμπεράσματά του και ε, όσον αφορά τις μελλοντικές πρωτοβουλίες προγραμματισμού το Συμβούλιο συμφωνεί με την ε, Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, μια κοινή προσπάθεια για την έρευνα αλλά δυστυχώς έχουμε μόνο μία δυνατότητα δηλαδή δια της των συμπερασμάτων του Συμβουλίου διότι η οδηγία μας δεν μας δίνει άλλη οικονομική ε, βάση. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Τώρα έρχονται οι ομιλητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων και καταρχήν η κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κύριε Πρόεδρε. Η Σουηδική Προεδρία θέλει το Δεκέμβριο να υθετήσει τα συμπεράσματά της σχετικά με την ε, καταπολέμηση αυτών των ασθενειών χωρίς να περιμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση πάνω στο θέμα αυτό και υποστηρίζω ένα ψήφισμα που θα ενστερνιζόταν τη θέση του Κοινοβουλίου όσον αφορά ε, την καταπολέμηση των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, κυρίω την όσο του Αλτσχάιμερ. Οι νευροεκφυλιστικέ ασθένειε είναι σημαντικό πρόβλημα υγεία στην Ευρώπη και ε, το επίπεδο ζωής σε ανεπτυγμένε χώρες οδήγησε σε μεγαλύτερη μακροζωία, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα περισσότερο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον αντίκτυπο, τις συνέπειες που έχει αυτή η ασθένεια όσον αφορά ε, εκείνους που περιθάλπτουν τους ε, ε ασθενείς. Είναι ένα πρόβλημα που θέτει σε δύσκολη θέση όλα τα συστήματα ε, περίθαλψης και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζεται σε πτυχές που αφορούν την έρευνα και το ψήφισμα που προτείνουμε εμείς ε, τονίζει και την, ε, ότι χρειάζεται υποστήριξη έρευνα και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνα θα βελτιώσει την κατάσταση. Λοιπόν, απευθύνω έκκληση. Α εστιάσουμε τι προσπάθειέ μα και στην επιστημονική έρευνα και στον τρόπο με τον οποίο αυτή η έρευνα αντικατοπτρίζεται στη φροντίδα των ασθενών δοθέντος του συμφέροντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα και τη σημασία που έχει το θέμα αυτό, ε, που είναι πιλωτικό πρόγραμμα για τον κοινό προγραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων, είναι ουσιώδες η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου να ληφθεί υπόψη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Υπενθυμίζω το άρθρο 182 ε, τη συνθήκη της Αβώνας που εξασφαλίζει τη νομική βάση για αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πατρίτσια Τόγια τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρωτοβουλία που συζητούμε είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον για την έρευνα, για την καταπολέμηση των ευρωεκφυλιστικών ασθενειών θα είχαμε προτιμήσει και το είχαμε πει μια πιο άμεση συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πολιτικό πρόγραμμα. Αν δεν θέλουμε να σταματήσουν τα πράγματα και θέλουμε να συνεχίσουμε, θα πρέπει να έχουμε εχέγγυα ότι η άποψή μα θα ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα και ότι θα διευκρινιστεί για το μέλλον μια πιο βέβαιη νομική βάση για μια πιο μεγάλη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό τη έρευνα. Πρέπει να παρέμβουμε όμω με απαραίτητα μέσα και πόρου ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε μια τόσο διαδεδομένη ασθένεια όπως ε, το Αλτσχάιμερ και άλλες παρόμοιες όπου δεδομένης της γύρανσης του πληθυσμού θα αυξηθούν στο μέλλον. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε μεγάλα προγράμματα ευρείας κλίμακος και για τη διάγνωση αλλά και για τον καθορισμό των θεραπείων. Θεμελιώδους είναι ε, ε, σημασίας η έγκαιρη διάγνωση, η πολυτομιακή προσέγγιση οι βάσεις δεδομένων, τα θεραπευτικά φάρμακα και αγωγές και τα μοντέλα θεραπείας που να είναι κατάλληλα και βεβαίως η παροχή υπηρεσιών που να είναι κατάλληλη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να γνωρίσουμε ούτε την ε, κοινωνική πτυχή των ασθενών, ούτε την συμμετοχή των ενώσεων ε, και οργανώσεων των ε, ασθενών και των συγγενών για την κοινή έρευνα θα πρέπει να, είμαστε, να επικεντρωθούμε και μέσα και πόρους, να αποφύγουμε επικαλύψεις, κατακαιρματισμούς και έτσι να φτάσουμε σε μια κρίσιμη μάζα που θα μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε εις ό,τι αφορά την έρευνα. Σε άλλες περιοχές του κόσμου, δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κοινού δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ επενδύων, κάτι το οποίο μας κάνει να κατανοούμε πόσα ακόμα πράγματα πρέπει να κάνουμε και μάλιστα επιγόντως σε κοινά προγράμματα, σε στατικές γραμμές, σε προγράμματα που να ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Κοινά προγράμματα μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, χωρίς να αγνοούμε τη διεθνή πτυχή του θέματος που, μπορέσει, θα μπορέσει να αποτελέσει μια κοινή πλατφόρμα σε διεθνές επίπεδο. Köszönöm, asszonyom. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό κατόπιν ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου. Σήμερα συζητάμε μια πρόταση ψηφίσματος για τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Κανονικά έπρεπε να είναι οδηγία και την επόμενη φορά πρέπει να συζητήσουμε οδηγία. Συμπεριλαμβάνουν εκτός από την Alzheimer και την Parkinson. Πρόκειται για ασθένειες που αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη. Το κόστος μακροπρόθεσμα θα αυξηθεί και πρέπει να γίνει πολλή έρευνα. Δυστυχώ υπάρχει πολλή διπλή έρευνα, πολλή γραφειοκρατία στην Ευρώπη. Γι' αυτό με την πρόταση ψηφίσματο θέλουμε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό αυτών. Η Γκουε κατέθεσε μία τροπολογία ε, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ καλή, δυστυχώ είναι λίγο λανθασμένη διατύπωση. Γι' αυτό ζητάω να αναδιατυπωθεί για να είναι καλύτερη η ρύθμιση. Υπάρχει ένα πρόβλημα πραγματικό με τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνία και θα ήθελα η Κομισιόν και το Συμβούλια να δουν το ζήτημα των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία στα φάρμακα, στα βιολογικά ζητήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι αρρώστιε. Εμεί, εν πάση περιπτώσει, υποστηρίζουμε αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλίπ Λαμπέρτς κατόπιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε. Αισθάνομαι λίγο απογοητευμένος ε, όσον αφορά τον εισηγητή σε αυτό το ψήφισμα. Τέλος πάντων δεν είναι τώρα η ώρα να μιλήσουμε για τα θεσμικά ζητήματα. Πρέπει να κινηθεί το Συμβούλιο. Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Πράγματι ελπίζουμε το Συμβούλιο να δεχτεί τις ιδέες που περιέχονται σε αυτό το ψήφισμα που θα ψηφιστεί αύριο. Πρέπει να περάσουμε σε μια σωστή ισορροπία μεταξύ, πώς λέμε, για προσαρμογή και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και εδώ πέρα πρέπει να έχουμε μια ισορροπία για να προλάβουμε αυτά τα φαινόμενα γιατί είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος να καταπολεμήσουμε την ασθένεια είναι λοιπόν αυτή η κοινή προγραμματική πρωτοβουλία αρκετή. Ε, καταρχήν πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα σε τέτοια μεγάλα εγχειρήματα η συνεργασία και να μην είναι κάτι το εθελοντικό, να είναι κάτι το δεσμευτικό για όλα τα κράτη-μέλη να αναγκαστούν να συνεργαστούν και κατόπιν όσον αφορά τις μουσιονομικές προτεραιότητες. Το πρώτο ερώτημα είναι εάν ξοδεύουμε αρκετά σε αυτές τις ασθένειες. Εμείς θεωρούμε ότι δεν γίνεται αυτό και θα ενθαρρύναμε στα επόμενα ερευνητικά προγράμματα να φύγουν λεφτά από μεγάλα προγράμματα όπως το ITER που μας λένε οι επιστήμονες ότι θα αποδώσουν σε 60 χρόνια και να πάνε κάποια από αυτά τα χρήματα στην έρευνα περί Αλτσχάιμερ και παρομοίων ασθενειών. Αυτό νομίζω χρειάζεται. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίζα Ματίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη μου υποστήριξη σε αυτά που είπε ο κύριος Ροέλ και ε, το βασικό πολιτικό ζήτημα που βρίσκεται εδώ ως διακύβευμα ή ο κοινό προγραμματισμός για την έρευνα. Αυτό το οποίο έγινε στα πλαίσια του κοινού προγραμματισμού για ε, την όσο Αλτσχάιμερ ήταν ότι στη μέση της διαδικασίας άλλαξαν οι κανόνες από έκθεση περάσαμε σε ψήφισμα, οπότε μειώθηκε η δυνατότητά μας στα πλαίσια της συναπόφασης να επηρεάσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό θα ήθελα να γνωρίζω αν τουλάχιστον αυτό το οποίο συστήνουμε, αυτό το οποίο προτείνουμε θα ληφθεί υπόψη όχι. Ο προγραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε θέμα είναι μια πολιτική και όχι μια τεχνική επιλογή. Από αυτή την έννοια ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω είναι πολιτική προτεραιότητα, όπου σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διαφανείς, πρακτικές και αποτελεσματικές. Αυτό το οποίο έγινε με τη διαδικασία σε σχέση με την κοινή απόφαση και τον κοινό προγραμματισμό της έρευνας για την ε, νόσο Αλτσχάιμερ είναι μια διαδικασία που δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθεί. Και αν τουλάχιστον παρατηρηθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον, παρακαλώ να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως για να λάβουμε τα μέτρα μας. Είναι θέμα που αφορά την ίδια την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Κατόπιν κυρία Ντότς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην εκλογική μου περιφέρεια στη Βόρεια Ιρλανδία έχουμε 16.000 ασθενείς από άνοια. Αυτοί και οι οικογένειές τους καθώς και οι θεραπευτές τους χρειάζονται μια πιο ενεργή αντιμετώπιση για να θεραπεύσουν αυτή την ασθένεια όσο γίνεται. Χρειάζεται λοιπόν πανευρωπαϊκή συνεργασία και πιστεύω ότι μια συνδυασμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση της ασθένειας μπορεί να μας δώσει νέα στοιχεία, νέες ανακαλύψεις και ίσως και νέα θεραπείες και φάρμακα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε περίπου 400.000 ασθενείς με Αλτσχάιμερ και μέχρι το 2025 μπορεί να φτάσουν αυτοί τις 750.000. Χρειάζονται λοιπόν έγκαιρες διαγνώσεις αλλά και περισσότερη κοινωνική έρευνα ιδίως για τις οικογένειες που εργάζονται ως θεραπευτές, οικογένειες θεραπευτών για να ληφθεί υπόψη η ζωή σε όλες τις, τις μορφές. Ευχαριστώ Περνάμε τώρα στους υπόλοιπους ομιλητές. Πρώτη έχει τον λόγο η κυρία Καρβάλιο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δηλώ την ικανοποίησή μου με τις δραστηριότητε που ανελήθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της καταπολέμησης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και ιδιαίτερα του Αλτσχάιμερ. Τα κρατημέλη έχουν κάνει ε, πολύ σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες. Είναι όμως σημαντικό η συνεργασία με τον, των κατών μελών να ενισχυθεί γιατί αυτό διασφαλίζει μεγαλύτερο συντονισμό στον τομέα της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής κινητικότητας και ε, έτσι αποφεύγουμε τον κατακαιρματισμό των ενεργειών μας. Οι ερευνητικέ δραστηριότητες ε, αποτελούν πολύ σημαντικό μέσα για τη μείωση του καταρκηματισμού αυτού και για να συμμετέχουν όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κρατημέλη, ιδιωτικό, δημόσιο ε, τομέα. Κοινό προγραμματισμό λοιπόν είναι κάτι που θα αποτελέσει κλειδί για το μέλλον του ευρωπαϊκού ερευνητικού χώρου. Η οικοδόμηση του οποίου είναι στο κέντρο τη ερευνητική πολιτική, τη πολιτική έρευνας, σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Κα... Εκφράζω λοιπόν την ανησυχία μου σε ό,τι αφορά τι εξελίξει για τον κοινό προγραμματισμό γραφειοκρατία, καθυστερήσεις, διοικητικά προβλήματα. Ερωτώ λοιπόν, τι προτιθέμεθα να κάνουμε για την οικονομία κλίμακος ε, ε, που θα πρέπει να εφαρμοστεί σε σεβασμό όλων της των πτυχών. Ανταγωνιστικότητα, σεβασμός του πλέον αδύναμου, κοινό προγραμματισμός που σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι κάτι που για τον τομέα είναι απολύτως απαραίτητο. Vielen Dank. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Τσέλντερς, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ως ε, επαγγελματίας στον τομέα της υγείας επί 30 έτη απογοητεύτηκα για όταν άκουσα πως το Κοινοβούλιο δεν θα παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση αυτή. Παρ' όλα αυτά πρέπει να προχωρήσουμε. Η κρίση αυτή βαθαίνει. Ο αριθμός ε, των κρουσμάτων παγκοσμίω θα πάει από τα 35 εκατομμύρια σήμερα στα 107 εκατομμύρια το 2050 και μία από τις ε, φρικτές συνέπειες είναι πως επηρεάζονται και άλλοι πλήν του ασθενή. Π.χ. στην Ιρλανδία υπάρχουν 5.000 εγγεγραμμένοι θεραπευτές που φροντίζουν ε, τους ασθενείς και αυτή η ασθένεια λέγεται και οικογενειακή ασθένεια γιατί βεβαίως αναγκάζεται όλη η οικογένεια να φροντίζει τον ασθενή. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην καταπολέμηση του Αλτσχάιμερ δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και η νέα κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβει είναι τη μοναδική συνεισφορά του Κοινοβουλίου και να βοηθήσει όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τους πάρα πολλούς ανθρώπους που τους φροντίζουν για να αυξηθεί η ποιότητα ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην διαδικασία Catch the Eye. Ζήτησαν τον λόγο κάποιοι ομιλητές. Πρώτα απ' όλα η κυρία Μαγκίνες έχει τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνδυασμό τη έρευνα σε αυτό το τομέα είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό προφανώ και δεν αφορά μόνο την ασθένεια του Αλτσχάιμερ αλλά όλε τι νευροεκφυλιστικέ ασθένειε. Το κοινοβούλιο μα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η έρευνα. Οι συνεννοήσεις με το Συμβούλιο για το θέμα παραδείγματος χάρη της εφημερίας των ζώων στα πειράματα ήταν αποτελεσματικές και ελπίζω να συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στην έρευνα, την έρευνα με ζώα ίσως με τρόπο πιο ανθρώπινο για τα ζώα αλλά είναι ακόμη απαραίτητο για να μπορούν να θεραπευτούν να βρεθούν θεραπείες για ανθρώπους μεταξύ των οποίων μπορεί να βρεθούμε και εμείς. Ελπίζω να υπάρξει στη δεύτερη ανάγνωση έγκριση της σημαντικής αυτής οδηγίας και αν και δεν υπέξαμε σημαντικό ρόλο εμείς μέχρι τώρα νομίζω ότι στο εξής θα το πράξουμε. Ευχαριστώ κατόπιν Σόνικ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα της ε, καταπολέμησης της ασθένειας ε, τέθη επί Γαλλικής Προεδρίας και πρέπει να είμαστε ευτυχείς γι' αυτό. Τότε υπόθηκε πως πρέπει να αναλυφθεί ευρωπαϊκή δράση και καλό θα ήταν να το δούμε με μεγάλη σοβαρότητα και οι επόμενες ε, προεδρίες. Ήδη ακούστηκε πως επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και τις οικογένειές τους που υποφέρουν μαζί τους. Όταν συναντάμε τους ε, ψηφοφόρους μας, ε, μας ρωτάνε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ρόλο παίζετε, γιατί πράγμα είστε υπεύθυνοι τέτοια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν για να οικοδομήσουμε και την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα λοιπόν των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Χουντής, κατόπιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ το πρόβλημα της καταπολέμησης των νευροεκφελιστικών ασθενειών και ιδιαίτερα του Αλσχάιμερ πάρα πολύ σοβαρό επομένω είναι πολύ χρήσιμο να υπάρξει και να επιτευχθεί συντονισμό των ενεργειών των χωρών τη ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αιτίε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρόληψης, της θεραπείας αλλά και των συνεπειών που έχουν τέτοιε νόσοι και στους ασθενείς και στο ευρύτερο δημόσιο σύνολο και στη δημόσια υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι η προτεραιότητα και η κύρια κατεύθυνση πρέπει να είναι στον τομέα της πρόληψης και όχι της φαρμακευτικής αγωγής ε, επίσης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κέντρα παρακολούθησης των ασθενών και των ατόμων που τους ε, φροντίζουν και όλο αυτό να εξασφαλίσει την ισότιμη επιστημονική συμμετοχή των κρατών στην ερευνητική αυτή προσπάθεια της ευρωπαϊκής ένωσης. τέλος αυτά τα δεδομένα που θα δημιουργήσει η βάση σε συνεννόηση του συμβουλίου και των μελών κρατών πρέπει να είναι κάτω από η δημόσια και κρατική ιδιοκτησία μέσα στα πλαίσια των εθνικών συστημάτων τα συμπεράσματα να ανακοινώνονται σε δημόσια φόρουμ παγκόσμια και ε, από εμά εξαρτάται να ελέγξουμε αυτόν τον προπολογισμό για το σχετικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δύο μιλητέ έχουμε ακόμα. Η κυρία για ένα λεπτό παρακαλώ. E, Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δώσουμε όση προσοχή, περισσότερη προσοχή γίνεται στην έρευνα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς του Αλτσχάιμερ. Έχουμε 27 χώρες μέλη και το καθένα δεν μπορεί από μόνο του να βοηθήσει τους ασθενείς. Γιατί τα υγειονομικά συστήματα, τα συστήματα περίθαλψης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και οι πόροι των χωρών διαφέρουν μεταξύ τους. Γι' αυτό επειδή πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη και το ότι και η οικογενειακή κατάσταση των ασθενών είναι πολύ διαφορετική μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει οπωσδήποτε συντονισμός και συνδυασμός των προσπαθειών πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση της έρευνας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει πραγματική βοήθεια των ασθενών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίος, κύριο Ρόλ, για ένα λεπτό. Äh, θα είμαι σύντομος, ε, κυρία Πρόεδρε. Το ανέφεραν πάρα πολλοί ομιλητέ πω υπάρχει μεγάλη ανάγκη να δράσουμε σε αυτόν τον τομέα. Πρόκειται για μια αρρώστια που αγγίζει όλο και περισσότερου ανθρώπου. Πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη, να ενώσουμε τι δυνάμει μα. Οπότε είναι λογική η οδός που ακολουθείτε εδώ πέρα. Κρίμα είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και τελευταία στιγμή αναγκάζεται να παρέμβει με ένα ψήφισμα το Κοινοβούλιο Λυπήρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικότερο είναι να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτοί ήταν ε, και οι τελευταίοι ομιλητέ από τη διαδικασία και τη ΕΕ. Τώρα το λόγο έχει το Συμβούλιο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το Αλτσχάιμερ και οι παρόμοιες ε, ασθένειες είναι πράγματι φρικτές αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει με στην οικογένειά τους το να προσβάλλεται κάποιος από μια τέτοια ασθένεια και βλέπουν τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο θέλουν οπωσδήποτε περισσότερη έρευνα στον τομέα αυτών. Πρέπει εδώ πέρα να συντονίσουμε καλύτερα την ε, έρευνα στην Ευρώπη το ευρωπαϊκό πιλωτικό σχέδιο λοιπόν είναι να χρησιμοποιηθούν οι καλύτεροι ευρωπαίοι ερευνητές για να συνεχίσουμε να ερευνούμε τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Υπάρχει λοιπόν συνεργασία μεταξύ της Γαλλίας, της Τσεχίας και της Σουηδίας και έχουμε ήδη αναγνωρίσει την σημασία του Αλτσχάιμερ σε σχέση με τη δημόσια υγεία Ήδη επί Γαλλικής Προεδρίας είχε γίνει μια σημαντική διάσκεψη και τον Σεπτέμβριο και η Σουηδική Προεδρία διοργάνωσε ένα συνέδριο με θέμα αξιοπρεπή γεράματα. Όπως ε, είπαμε θα καταλήξει το Συμβούλιο σε συμπεράσματα στις 3 ε, Δεκεμβρίου και οπωσδήποτε θα ληφθεί υπόψη το αυριανό σας ψήφισμα το ζήτημα του Αλτσχάιμερ θα επανέρχεται οπωσδήποτε και στα επόμενα προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λέει και η Πρόεδρος τελείωσε η συζήτηση για αυτό το ζήτημα. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Σύμφωνα λοιπόν με την ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα τις παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 150 του κανονισμού. Να ξεκαθαρίσω από τώρα πως υπάρχουν πολύ περισσότερες ερωτήσεις από τον χρόνο που έχουμε